Um, Συνάδελφοι, ξεκινάμε με τις ανακοινώσεις της Προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών σήμερα το πρωί. Εξετάσαμε θέματα γύρω από τις νομοδοτήσεις που πρέπει να ετοιμάσουμε και οι συντονιστές συνιστούν να υπάρξει μια γνωμοδότηση για την μεταφορά στο Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. We agree also that on the motion for του λεγόμενου πρωτοδικίου. Τώρα σχετικά με την πρόταση του κυρίου Μπονάνο για το πρόγραμμα το ετήσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπαμε ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια σε επίπεδο δικής μας Επιτροπής γιατί τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο έτος αντιμετωπίζονται από τις πολιτικές ομάδες σε αυτή τη φάση και το ψήφισμα στην Ολομέλεια περνάει μέσα από τις πολιτικές ομάδες και όχι από τις επιτροπές. Δεν μπορούμε φυσικά να βοηθήσουμε τον κύριο Μπονάνο, αλλά μπορεί μέσω της πολιτικής του ομάδας αν θέλει να κάνει πρόταση για την απόρριψη του προγράμματος της Επιτροπής. Τώρα, πρόταση ψηφίσματος που ζητά από τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θέματα όλα αυτά βέβαια που άπτονται εθνικών αρμοδιοτήτων και δεν έχουμε κάτι να κάνουμε εμείς σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σχετικά τώρα με την ηλεκτρονική δημοκρατία, το e-democracy. Θα υπάρξει ακρόαση 15 και 16 Μαρτίου. Η ΑΦΚΟ δέχεται την πρόταση της ΛΥΜΠΕ να υπάρξει μια κοινή ακρόαση το μήνα Φεβρουάριο στα πλαίσια του μηχανισμού για τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Ο Σέφλινγκ είναι εισηγητής επί τη βάση του κανόνα 53 συν, βελτιωμένου δηλαδή, και υπήρχε μια συμφωνία ανάμεσα στους δύο Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε. Συμφωνήσαμε επίσης ότι η μέρα επίσκεψης στην ΑΦΚΟ προσκαλούνται όλα τα μέλη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο στις 17 Φεβρουαρίου του 2016. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια και από την στάση του δικαστηρίου. Εμείς έχουμε πρόβλημα με τις ημερομηνίες μέχρι τώρα, όχι αυτή. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι επίσης ανακοινώσεις δικές μου. Ήμουν εκπρόεδρος των αντιπροσωπιών μας στη Ουάσιγκτον και στο Λονδίνο τον μήνα Νοέμβριο. Θα ξεκινήσω σύντομα με την αποστολή στο Ουάσιγκτον. Είχαμε μια μεγάλη αντιπροσωπεία με πολλές πολιτικές ομάδες. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη η ΑΦΚΟ, η οποία δεν είναι τομεακή επιτροπή. Ξέρετε ότι αλλιώς οργανώνονται οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο ε, Κογκρέσο, ανάλογα με τομείς της οικονομίας ή της πολιτικής. Έτσι λοιπόν καταφέραμε να αποδείξουμε μέσα από την επίσκεψη αυτή και τις συναντήσεις μας ότι αυτό το οποίο έχει σημασία στα πλαίσια της ατζέντα αυτής είναι οι αξίες, οι ομοιότητες και οι διαφορές σε επίπεδο αξιών από τις οποίες πολλά μπορούμε να μάθουμε. Το δεύτερο θέμα που θέλω να υπογραμμίσω για το μέλλον είναι ότι συνήθως παραπονούμεθα στο Κοινοβούλιο ότι σχετικά με τη Washington δημιουργείται μια κατάσταση σύμφωνα με την οποία υπάρχουν πολλές αντιπροσωπείες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πηγαίνουν ταυτόχρονα στο Κογκρέσο και αυτό δεν είναι καλό. Εγώ νομίζω ότι είναι καλό. Αυτή η ισχυρή παρουσία διαφορετικών αντιπροσωπιών ταυτόχρονα νομίζω ότι δημιουργεί μια κριτική μάζα της παρουσίας που τονώνει το βάρος, αυξάνει το βάρος της παρουσίας μας εκεί και το ενδιαφέρον α, της, για την επίσκεψή μας στα αμερικανικά θεσμικά όργανα. Νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερες κοινέ συνεδριάσεις πριν πάμε εκεί και αφού πάμε εκεί, γιατί υπάρχει παρόμοιο ενδιαφέρον για πάρα πολλά θέματα και νομίζω ότι η επόμενη συνάντηση όταν γίνει ε, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται και από περισσότερες κοινέ συνεδριάσεις. Θα ήθελα να υπογραμμίσω και κάποια άλλα θέματα, γιατί η επίσκεψη αυτή ήταν πολύ καλή. Είχαμε συναντήσεις με πάρα πολλές αμερικανικές υπηρεσίες, εκπροσώπους όλων των κυβερνήσεων, think, των, της κυβέρνησης μάλλον, υπηρεσιών, think tanks, και ίσως να επανέλθω σε αυτά λίγο σε λίγο. Νομίζω ότι μπορούσαμε να συναντήσουμε ένα φάσμα μεγάλο των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για διάφορους τομείς και ήταν πολύ σημαντικό αυτό για μας. Πήγαμε εμείς εκεί σε μια περίοδο που υπήρχε ένταση ανάμεσα στο Κογκρέσο από τη μία και την κυβέρνηση από την άλλη. βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο η οποία ονομάζεται της διχασμένης κυβέρνησης και η διαδικασία αυτή για μας ήταν πηγή γνώσης. Ήμασταν επίσης εκεί σε μια περίοδο που είχε ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία για την Προεδρία. Είχαμε μια συνάντηση με τον διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας της Χίλαρη Κλίντον και ενημερωθήκαμε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διαδικασία αυτή. Και αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι μπορέσαμε να δούμε τι σχέσεις υπάρχουν ανάμεσα στο κεντρικό επίπεδο και στο περιφερειακό επίπεδο. Πήγαμε στο Μέριλαντ και σε άλλες περιοχές, είδαμε το σύστημα ελέγχου ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα, από το ομοσπονδιακό, από το κεντρικό κρατικό, τις σχέσεις ανάμεσα στις πολιτείες, και νομίζω ότι συναντήσαμε και εμπειρογνώμονες οι οποίοι ε, γνωρίζουν πώς δουλεύει το σύστημα αυτό και το είχαμε ανάγκη. Υπάρχουν πολλά μαθήματα για την Ευρώπη ακριβώς στα πλαίσια των λύθεων, τις οποίες ε, είδαμε να έχουν ε, δημιουργήσει, να έχουν βρει οι Αμερικανοί. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, στα πλαίσια της ΑΦΚΟ είδαμε πώς λειτουργεί το Κογκρέσο σε σχέση με διαφάνεια, κώδικα συμπεριφοράς η Επιτροπή Δεοντολογίας, επισκεφθήκαμε το κέντρο έρευνας, ζηλέψαμε πάρα πολύ εκεί για την τεράστια δυνατότητα που έχει το κέντρο τεκμηρίωσης του Αμερικανικού Κογκρέσου με πάρα πολλούς εργαζομένους και σκεφτήκαμε ότι πραγματικά θα έπρεπε να δημιουργήσουμε κάτι αντίστοιχο και παράλληλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι βρισκόμαστε αιώνες πίσω από την ικανότητα την οποία έχουν οι Αμερικανοί να στηρίζουν και να τεκμηριώνουν μέσω της έρευνάς τους στην καθημερινή τους δουλειά. Τελειώνοντας την επόμενη φορά που θα πάμε, θα πρέπει νομίζω να έχουμε ένα στενότερο πρόγραμμα, λιγότερους στόχους. Ενδιαφέρουσα αυτή η οριζόντια συζήτηση, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να την κάνουμε καλύτερα συγκεντρώνοντας σε λιγότερα θέματα. Νομίζω επίσης ότι κάναμε όμως πολλές επαφές, προσκαλέσαμε πολλούς, ε, πολλά μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, ακόμα και τη Rachel Stapp, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαπραγμάτευση στα πλαίσια του TTIP. Υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας με τους Αμερικανούς για να δούμε πώς μπορούμε να ωφεληθούμε από τη συνεργασία όχι μόνο σε τομιακό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο διακανονιστικό. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφοι που ήταν στι Ηνωμένε Πολιτείε. Περνάμε τώρα, γενικά πάω γρήγορα βέβαια. ο Σέφλιν. Σύντομα, είπε τα πάντα περίπου. Ένα από τα θέματα τα οποία εμένα μου μείναμε είναι ότι το Κογκρέσο λειτουργεί εντελώς διαφορετικά σε επίπεδο νομοθετικό από ό,τι εμείς εδώ. Νομίζω ότι υπάρχει με ένα δικοματικό σύστημα, αλλά στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και βεβαίως <clears throat> είναι σημαντικό να δει κανεί ότι υπάρχουν πολύ έντονες διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των κομμάτων και ότι οι σχέσεις μεταξύ ρεπουμπλικάνων και δημοκρατικών δεν είναι σε καθόλου, καθόλου καλά επίπεδα. Χειρότερα παρά ποτέ. Είδαμε επίσης ότι ουσιαστικά οι σχέσεις που έχουμε εμείς εδώ με τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν μπορούν καθόλου να παρομοιαστούν με τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ της Ομοσπονδιακής και της ε, και των αρχών των πολιτιών. Καμία σχέση. Εμείς πήγαμε όντως στο Μέριλανδ και ακούσαμε τη συζήτηση που λαμβάνει η χώρα εκεί και για την ανεξαρτησία των ε, αρχών των διαφόρων πολιτιών. Καμία σχέση με αυτά που συζητάμε εμείς εδώ. Πρόεδρος. Συναντηθήκαμε επίσης και με ειδικού για θέματα ε, κομμάτων, ε, για την, τους υπεύθυνους για το δικοματικό σύστημα. Και συναντήσαμε και δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους. Όντως δεν υπάρχει καλή συνεργασία, καλές επαφές και οι εκπρόσωποι τους και σε θέματα που αφορούν ε, το Λευκό Οίκο αλλά και το Κογκρέσο Όπως ξέρετε είδαμε και κάποιους ε, από πανεπιστήμια που ασχολούνται με την ευρωπαϊκή πολιτική. Υπάρχει μάλιστα και μια έδρα ζωμονέ σε ένα από τα πανεπιστήμια τους. Πιστεύουμε ότι όσον αφορά τουλάχιστον την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επαφές, η κατανόηση που έχουν για την ευρωπαϊκή πολιτική είναι βεβαίως μεγαλύτερη από αυτή της δυτικής ακτής. Αλλά παρόλα αυτά σίγουρα θα πρέπει οι επαφές να εντατικοποιηθούν. Τώρα, το δεύτερο ταξίδι, η δεύτερη αποστολή στο Λονδίνο με πολλούς συναδέλφους θα σας αφήσω να πάρετε το λόγο εσείς. George, ξέρω ότι φεύγεις, οπότε σκοπός μου είναι να ακούσουμε και κάποιον άλλο. Πώς έχουν τα πράγματα στο Λονδίνο λίγους μήνες πριν το δημοψήφισμα. Ευχαριστώ. Όχι, εγώ δεν θα σας παρουσιάσω τώρα το Λονδίνο, αλλά τις εντυπώσεις μου Όλοι γνωρίζετε ότι υπάρχουν τα τέσσερα σημεία του David Cameron στην αποστολή που έστειλε στον Donald Tusk. Η γενική μου εντύπωση είναι ότι μακροπρόθεσμα, ό,τι και να συμβεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να Πήγα να ότι μέχρι το Δεκέμβριο τη Σύνοδο Κορυφής θα έχουν υλοποιηθεί, θα έχουν επεξεργαστεί όλα αυτά τα σημεία. Αυτό σίγουρα μπορεί να επηρεάσει και την ημερομηνία του δημοψηφίσματος. Εάν βεβαίως ε, ακούσουμε κάποιες θετικές, υποστηρικτικές προτάσεις ότι ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Συγγνώμη Ρίτσαρτ, θα επανέλθω θα μπορούσε να γίνει ταχύτατα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν θα προλάβουν τόσο γρήγορα. Είχα μια σχετικά, ε, πολύ θετική εντύπωση της Χίλερη Μπέν και τη Πατ Μακάρτη από το Εργατικό Κόμμα τις προτάσεις τους για τα κοινωνικά θέματα καθώς και των τον αρμόδιο των εργατικών για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. Ακούσαμε τις προτάσεις τους. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι το θέμα των επιδομάτων, ε, οικογενειακών επιδομάτων που στέλνονται από μετανάστες, ευρωπαϊκές χώρες, τις χώρες προέλευσής τους. Περίπου μία ώρα κάτσαμε τον Άλεξ Άλμον από το Εθνικό Κόμμα της Σκοτίας. Στη Σκοτία, τουλάχιστον αυτό κατάλαβα, είναι περίπου 60% υπέρ του να παραμείνει η Μεγάλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 40% κατά. Σαφέστατα υπέρ λοιπόν. Και από ό,τι καταλάβαμε, ε, εκείνοι τουλάχιστον δεν πρόκειται να συνεργαστούν με άλλες πολιτικές δυνάμεις, πολιτικά κόμματα. Αυτό βεβαίως, αν θέλετε, είναι τελείως διαφορετικό με αυτό που συνέβη το 1975 όπου τα τρία μεγάλα κόμματα, δηλαδή τα δύο μεγάλα κόμματα και οι φιλελεύθεροι συνεργάστηκαν. Οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, μας είπαν ότι έχουμε μάθει πολλά, έχουμε διδαχτεί πολλά από το δημοψήφισμα στην Σκοτία. Εγώ προσωπικά έχω την εντύπωση ότι αυτοί που θέλουν να φύγει η Μεγάλη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μια πιο ελκυστική ιστορία να διηγηθούν. Το μήνυμά τους είναι ίσως πιο εντυπωσιακό, έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο, συναισθηματικό αντίκτυπο και αυτό βεβαίως κατά την άποψή μας θα έχει ανητικές συνέπειες και για τη Μεγάλη Βρετανία γιατί θα υπάρξει μεγάλος διαχωρισμός αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βόρεια Ιρλανδία τώρα. Αν προχωρήσει το Brexit θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και με την Βόρεια Ιρλανδία και την ειρνευτική διαδικασία και δεν ξέρω αν ο ε, ε, Ρίτσαρτ ε, θα συμφωνήσει μαζί μου. Ο Γιολάινεν έχει όμως πρώτο το λόγο. Ναι. Βεβαίως υπάρχει κατάλογος ομιλητών και υπάρχει μια σειρά. Yeah, Ο Ρίτσαρτ Εγώ πήγα στο Λονδίνο και συμφωνώ με τον κύριο Σέπλιν ότι είναι πιο εντυπωσιακό το μήνυμα αυτών που είναι υπέρ του να βγει η Μεγάλη Βρετανία. Λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόνο αρνητικές πτυχές, μειονεκτήματα και βεβαίως Εμείς ρωτήσαμε πώς αυτά τα τέσσερα σημεία θα τα προωθήσει ο Κάμερον, πώς θα μπορέσει να τα πουλήσει στον κόσμο. Εγώ δεν έχω πραγματικά την εντύπωση ότι αυτά τα τέσσερα σημεία θα επηρεάσουν ε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό το δημοψήφισμα. Στο τέλος άλλα θα μετρήσουν και τα δημοψηφίσματα για την Ευρώπη όπως ξέρετε είναι παγίδες γιατί συνήθως οι ψηφοφόροι δεν απαντούν στα ερωτήματα που τίθενται. Απαντούν σε άλλα ερωτήματα τα οποία τους απασχολούν εκείνη την εποχή. Και έχω την εντύπωση ότι θα χρησιμοποιηθούν απλά μηνύματα από εδώ και πέρα στην προεκλογική εκστρατεία θα πούνε δηλαδή γιατί, και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί παραδείγματο χάρη είναι σημαντικό να παραμείνει η Μεγάλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω παραδείγματο χάρη αν αρχίσουμε να μιλάμε για την κόκκινη κάρτα, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσουμε κάποιους που ζουν στην ε, Βόρεια Ιρλανδία ότι αυτό θα έχει άμεσες επιπτώσεις και θα αλλάξει την καθημερινή του ζωής. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ενότητα και η ομάδα υπό, περί τον Πρωθυπουργό που πραγματικά προσπαθούν να προωθήσουν τα μηνύματα ενότητας θα ζητήσουν γραπτές διαβεβαιώσεις ότι είτε θα αλλάξει τώρα η συνθήκη είτε θα αλλάξει αργότερα. Αλλά θα θέλουν γραπτές διαβεβαιώσεις. Και επιθυμούν με ταχείες διαδικασίες και κεκλεισμένων των θερών να επιτευχθεί μια συμφωνία σε δύο εβδομάδες στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου. Εμείς όλοι βεβαίως Θέλουμε να δώσουμε κάτι στον David Cameron για να μπορέσει να γυρίσει σπίτι του στη χώρα του με κάτι απτό έτσι ώστε να μπορέσει η Μεγάλη Βρετανία να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θυμάμαι στο Στρασβούργο πριν από δύο εβδομάδες η Μαρίν Λεπέν, το Front National, είπε ότι αν πετύχουν οι Βρετανοί καλύτερες συνθήκες για την ε, Μεγάλη Βρετανία, εμείς όταν έρθουμε στην εξουσία θα ζητήσουμε καλύτερες συνθήκες για τη Γαλλία. Το ίδιο θα κάνουν και οι Πολωνοί και οι Ούγγροι και όλοι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι να γίνει καλύτερη Ευρώπη, καλύτερες συνθήκες για την Ευρώπη και όχι να επιλέγει η κάθε χώρα ότι βλέπει ότι μπορεί να αποφέρει ένα όφελος για την ίδια τη χώρα. Είναι σαφώς κάτι που θα πρέπει να το δούμε σφαιρικά, συνολικά. Είναι σημαντικό να δούμε τι μπορεί να μας ενώσει και όχι τι θα μας χωρίσει περισσότερο. Έχουμε την κυρία Diane James από την UKIP. Κυρία... Ε, σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να έρθω σήμερα και να θέσω ερωτήσεις. Ενδιαφέρθηκα από τις δύο προηγούμενες ομιλίες να πω ξεκαθαρίζοντας ότι είμαι θετική σε σχέση με τη δυνατότητα Brexit και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα και για μια καλύτερη Ευρώπη. Ε, νομίζω αυτό δεν ταυτίζεται με το κάτι καλύτερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιστολή του κυρίου Τάσκα στον Ντέιβιτ Κάμερον, της οποίας αντίγραφο έχω εδώ και μπορείτε να διαβάζετε, είναι ενημερωτική. Θέτει κάποια από τα σημεία τα οποία μας ενδιαφέρουν. Θα ήθελα λοιπόν κάποια σχόλια εδώ. Μιας και οι αλλαγές θα απαιτήσουν ξεκάθαρες και αδιαμφισβήτητες και ίσως και περίπλοκες αλλαγές στις συνθήκες. Θα διαφωνήσει κάποιος με τις προτάσεις αυτές. Πρώτον, το ερώτημα το οποίο θα πρέπει να τεθεί στην καλύτερη περίπτωση είναι μια υπόσχεση ότι κάπου κάποτε στο μέλλον οι συνθήκες θα αλλάξουν και θα έχουν νομική ισχύ οι αλλαγές αυτές. Δεύτερον, ότι οι διαδικασίες αυτές θα απαιτήσουν τη συμφωνία του Συμβουλίου σε ορισμένες περιπτώσεις και δημοψηφίσματα σε κράτη-μέλη, σε ορισμένα και επικύρωση από τα 28 κράτη-μέλη σύμφωνα με τις δικές τους συνταγματικές ρυθμίσεις. Επί της ουσίας τώρα. Το Brexit είναι στην ουσία ένα μικρό IOU σου οφείλω χωρίς ε, ημερομηνία, χωρίς νομικές δεσμεύσεις. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό είναι που θέλει να πετύχει το Ηνωμένο Βασίλειο. Δυστυχώς η πολιτική μας δεν είναι ειλικρινής και νομίζω ότι θα ήθελα να υπάρξει ειλικρίνεια από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ που ακούσατε τα σχόλιά μου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν κατάλαβα, μιλάμε ήδη για το ζήτημα της μαλευτανίας. ή τα κάνουμε όλα μαζί. Γι' αυτό δίσταζα να έγραφω στον κατάλογο. Να διευκρινίζω πως αρχικά προτείναμε δύο σημεία διότι ο Τζόναθαν ήθελε να έρθει αλλά δεν κατέστη δυνατόν. Γι' αυτό έγινε αυτό το μπλέξιμο. Ευχαριστώ. Και εγώ όπως ε, και άλλοι συνάδελφοι επέστρεψα λιγότερο αισιόδοξη με τη δυνατότητα να παραμείνει η, η Μεγάλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά αυτή την επίσκεψή μας στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Δόθηκε η εντύπωση ότι αυτό που ονομάζει ο Ρίτσορ Κόρβετ Brexit by accident, δηλαδή μια επιλογή που θα είναι το αποτέλεσμα μια σειράς γεγονότων ε, κακώς προγραμματισμένων. Αυτό το οποίο κατέστη σαφές από τη συζήτηση και με πρόσωπα σε υψηλές θέσεις ότι όλοι έχουν ήδη πάρει θέση για να μείνουν ή για να φύγουν ακόμα και σε επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών, προέδρων κοινοβουλευτικών επιτροπών και αξιωματούχοι υπεύθυνων κέντρων ερεύνας όλοι δηλώνουν ότι τους προσεχείς μήνες ή τουλάχιστον με σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ε, κατασταλάξουν ως εκ τούτου η διαδικασία που θα ξεκινήσει με τον Πρωθυπουργό στην ουσία χρησιμεύει στο να λάβει απόφαση ο ίδιος ο Πρωθυπουργό και να μεταθέσει αυτό που ορισμένοι μας είπαν ήδη ε, μερικές ε, μερικά εκατομμύρια ψήφων τουλάχιστον αυτά εγώ κατάλαβα από τις συναντήσεις που είχαμε στο Λονδίνο. Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά κάτι που ο Γιολάινεν ήδη ανέφερε ότι δηλαδή δεν μπορούμε να δεχθούμε την ιδέα μιας Ευρώπης ε, στην οποία υπάρχουν ε, χώρες οι οποίες επιθυμούν να ε, πάρουν όλο και περισσότερα κονδύλια για πάρτι τους. το πρόβλημα, το ζήτημα εδώ είναι να μείνουμε όλοι μαζί ενωμένοι και όχι κάποιος να πάρει παραπάνω από όλους τους άλλους. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να καταστρέψει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και θα οδηγήσει σε μια χειρότερη Ευρώπη, κάτι που ο Κάμερον δεν επιθυμεί. Διότι αναγνωρίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού σχεδιασμού και του ευρωπαϊκού οράματος. Ακριβώς λοιπόν επειδή αυτή, λοιπόν καταρχάς, αυτή η διαπραγμάτευση δεν μπορεί να διεξαχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, διότι αν χρειάζεται να είναι μια διαδικασία, κάτι με το οποίο εγώ δεν συμφωνώ, να χρησιμεύσει το να καθορίσει καλύτερα τις εγγυήσει για τα κράτη-μέλη προκειμένου να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περί αυτού πρόκειται στην ουσία Θέλω να είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν θα μου πάρει κάτι από το κράτος μου εκτός από έναν παγκόσμιο πόλεμο. Κανένα λοιπόν δεν θα μου αφαιρέσει κανένα κομματάκι εκτός από τη Ρωσία που θα μπορούσε να το κάνει. Είναι σαφές λοιπόν πως πρόκειται για επαναπροσδιορισμό και επανασυζήτηση του συμφώνου μας, του συμφώνου που μας ενώνει και να αξιολογήσουμε αν μπορούν να δοθούν να ε, γίνουν παραχωρήσεις όχι στη Μεγάλη Βρετανία αλλά αν μπορούν να γίνουν πράγματα παραπάνω στον βωμό της αυτονομίας ε, των επιμέρους κρατών. Θα δούμε μετά ποια θα είναι η πλειοψηφία η κατά. Για μια φορά, και καλή λοιπόν θα πρέπει όσοι κρίνουν ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο σοβασμός της ε, κυριαρχίας ή των εθνικών κυριαρχιών να δηλώσουν όλοι, όχι μόνο η Μεγάλη Βρετανία, να δηλώσουν λοιπόν τι προτίθενται να κάνουν, τι εννοούν με κάτι τέτοιο. Και συγκεκριμένα αυτό που ζητάει ο Κάμερον δεν είναι σοβαρό, αλλά το θέμα είναι πως όλο μαζί έχει ως αποτέλεσμα να αποδυναμώσει μια πολιτική Ευρώπη, μια Ευρώπη η οποία πηγαίνει προς ένα κοινό πολιτικό σχέδιο. Αν πρέπει να συζητηθεί το θέμα, θα πρέπει να συζητηθεί το πώς αυτή η ανησυχία που ε, έχουν πολλοί ότι τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να διαγραφούν από το κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο, τότε θα πρέπει να συζητηθεί, επαναλαμβάνω, αλλά για όλους και με όλους μέσα στα απαραίτητα χρονικά όρια και προθεσμίες και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλακεί άμεσα, αυτό δεν ενδιαφέρει φυσικά τον κύριο κάμερα, διότι είναι ως το εκλεγμένο όργανο των Ευρωπαίων πολιτών. Υπενθυμίζουμε ότι ε, τα κράτη εκπροσωπούν τους πολίτες τους, αλλά και εμείς κάνουμε το ίδιο. Η διαφορά είναι ότι εμείς εκπροσωπούμε όλους, δηλαδή ο Τζορ Κόρμπεθ και εγώ εκπροσωπούμε 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών περίπου πάνω κάτω ίσως λίγο παραπάνω, ενώ όποιος εκπροσωπεί το μεγαλύτερο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσωπεί τους πολίτες του και η πιο μεγάλη χώρα είναι η Γερμανία που η κυρία Μέρκελ δηλαδή εκπροσωπεί 70-80 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Όχι παραπάνω. No more. Αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε, το έχουμε κατά νου. Πρέπει να συζητάμε λοιπόν με στένος αυτά τα ζητήματα και φυσικά μπορεί να είναι νομικά δεσμευτικό και όταν αποφασίσουμε τι θα είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε και να παραχωρίζουμε θα χρειαστεί να ανοίξουμε τις συνθήκες, να τις αναθεωρήσουμε και μέσα στις συνθήκες να βάλουμε και άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται να δώσουμε μόνο μια απάντηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά να βάλουμε και πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν άλλα κράτη, αρνητικά κατ' εμέ, αλλά και θετικά ίσως. Θετικά αρνητικά πάντως, εξαρτώνται ανάλογα από την οπτική γωνία που τα βλέπει ο καθένας. Θεωρώ λοιπόν ότι κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί ότι αυτή η δικασία μπορεί να είναι ταχύτατη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήταν ενδιαφέρουσε συναντήσει στο Λονδίνο. Χαίρομαι που πολλοί συνάδελφοι πήραν είδηση του τι συμβαίνει εκεί. Και είδατε και διάφορες πλευρές της συζήτησης, τις οποίες από τις απλές ειδήσει στο παρελθόν δεν γνωρίζατε. Νομίζω όμως ότι χρειάζεται να το πλαισιώσουμε κάπως. Γιατί υπάρχει αυτό το δημοψήφισμα για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς έχει σχέση με την διαχείριση από που των βαθύτατων διαιρέσεων στο εσωτερικό του συντηρητικού κόμματος γύρω από την Ευρώπη. Είναι διαιρεμένοι σε πολύ μεγάλο βάθος και ο Πρωθυπουργός σαν ηγέτης του κόμματος είπε ότι πριν από τις ε, ε, εκλογές ότι μετά τις εκλογές εμείς θα προσπαθήσουμε να ε, βοηθήσουμε έτσι ώστε να αλλάξει προς το καλύτερο και να μεταρρυθμιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το είπε έτσι ώστε να μετριάσει τις διαφωνίες οι οποίες υπήρχαν στο εσωτερικό του κόμματός του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Ε, πολύ πιθανό ήταν να μην πίστευε το τι θα γινόταν μετά γιατί δεν ήξερε ότι θα μπορούσε να πετύχει μια απόλυτη πλειοψηφία και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να συζητήσει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια κυβέρνηση συνασπισμού με τους φιλελεύθερους δημοκράτες. Δεν πήγαν έτσι τα πράγματα. Δεν έχει νομίζω εξετάσει σε βάθος τι αιτήματα μεταρρυθμίσεων μπορεί να θέσει. Και νομίζω ότι έπρεπε να ψάξει για να βρει κάτι το οποίο μπορεί να είναι κάτι το συνηθισμένο αλλά και το που να μην είναι συνηθισμένο αλλά μην είναι και ανέφικτο. Δεν μπορεί να είναι ε, ανέφικτο βέβαια γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δεχτεί να τα συζητήσει, δεν μπορεί να είναι και ασήμαντο όμως. Και γι' αυτό έκανα αυτές τις τέσσερις προτάσεις που δεν ζητούν opt-out για το μη συγκεκριμένους ε, δεν λέει ότι θα πρέπει η Αγγλία να σταματήσει να συμμετέχει στην εφαρμογή διαφόρων πολιτικών. Δεν είναι αυτή η προσπάθειά του. Όλοι γνωρίζετε το πακέτο αυτό των τεσσάρων, το καλάθι των τεσσάρων. Και όπως είπε ο Λάινεν, αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν σημασία σε σχέση με το δημοψήφισμα. Ε, οι άνθρωποι θα αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν με βάση μόνο και μόνο τις επιμέρους μικρές ρυθμίσεις και νομίζω ότι η κυρία Τζόνς θα συμφωνήσει μαζί μου ότι το 90% δεν θα ασχοληθεί με λεπτομέρειες. Είναι όμως κρίσιμο για ένα 10 με 15% του εκλογικού σώματος, μεταξύ των οποίων και για τους κεντρώους του συντηρητικού κόμματος. Πρέπει να ζητήσει και να πετύχει κάτι το οποίο να φαίνεται αξιόπιστο, γιατί αυτό θα βοηθήσει το κοινό να τον στηρίξει. Ε, ίσως οι μεταρρυθμίσεις του να μην μας αρέσουν είτε σε επίπεδο ευρωπαϊκό, είτε σε επίπεδο εργατικού κόμματος, είτε άλλου κόμματος. Όμως το δημοψήφισμα δεν θα είναι ένα απλό ναι ή όχι στις μεταρρυθμίσεις. Το δημοψήφισμα είναι ναι ή όχι στην ευρύτερη εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα ή έξω και ίσως κάποιες τέτοιες μεταρρυθμίσεις να μπορούσαν να είναι αντιστρέψιμες, αλλά ένα μέσα ή έξω προφανώς δεν είναι κάτι το αναστρέψιμο. Πάντως είναι κρίσιμο λοιπόν να μπορέσει ο Κάμερον να δείξει ότι κάτι έχει πετύχει. Και μένα δεν θα μου αρέσει αυτό, αλλά πρέπει να έχει κάτι. Τώρα, πόσο δύσκολο είναι να το πετύχει αυτό. Αυτό θα εξαρτηθεί εν πολλής από τα μέσα τα οποία θα απαιτήσει. Παράδειγμα, κόκκινη κάρτα από ομάδα κοινοβουλίων. Θα μπορούσε να πει κανείς, πάρτε την υπάρχουσα διαδικασία με το όριο τη γίτρινη κάρτα, το όριο τη κόκκινη κάρτα, την πορτοκαλί συγγνώμη, και να πούμε στην Επιτροπή ότι αν φτάσουμε ας πούμε σε αυτό το επίπεδο τότε εμείς αυτόματα θα αποσύρουμε την πρόταση. Δεν πρόκειται να περάσει από το Συμβούλιο, οπότε θα πρέπει να σταματήσει αμέσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πορτοκαλί κάρτα. Αν όμως υπάρξει αίτημα για αλλαγή της συνθήκης ή του πρωτοκόλου του συνοδευτικού, αυτό είναι πρόβλημα γιατί θα απαιτήσει την επικύρωση από 28 κοινοβούλια. Και το αίτημα για την λεγόμενη ολοένα πιο εμβαθυμένη και ολοκληρωμένη ένωση. Σύμφωνα με τις αρχές της επικορικότητας βέβαια. Ο μύθος ε, του υπερσυγκεντρωτικού κράτους είναι ένας μύθος, δεν υπάρχει. Αλλά κάτι πρέπει να φέρει πίσω. Αν είναι μια δήλωση σύμφωνα με τις προτάσεις του Συμβουλίου της 24ης ε, 2014 ε, ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία λοιπά, τόσο το καλύτερο. Θα μπορούσε να συμφωνήσει ίσως κανείς. Αν επιμένει όμως να υπάρξει αναδιατύπωση της συνθήκης ή να υπάρξει ένα νέο συμπληρωματικό πρωτόκολλο, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όλα αυτά λοιπόν είναι υποσυζήτηση. Για το όριο τώρα των τεσσάρων ετών κάποιος ο οποίος με, τα πηγαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα την χάνει ε, των βοηθημάτων και της κοινωνικής κάλυψης αν δεν περάσουν τα τέσσερα πρώτα χρόνια. Αυτό είναι θέμα τεχνικό το οποίο πολλές φορές ισχύει και για τους ίδιους τους Βρετανούς και θα δημιουργήσει προβλήματα στην ίδια του τη χώρα ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρέπει να αλλάξει η κοινοτική νομοθεσία, οπότε αυτό θα πρέπει να περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή θα πρέπει να υπάρξει ένα πρωτόκολλο στη συνθήκη, μια τροπολογία στη συνθήκη. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είχε γίνει για την Ιρλανδία, για τη Δανία στο παρελθόν, είναι κάτι το εφικτό. Πάντως ο βαθμός δυσκολίας κάθε φορά με όλα αυτά τα επιμέρους θέματα αυξάνεται και δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της διαδικασίας. Κανένας δεν θα ήθελε να προκαλέσει σε ένα άλλο κράτος μέλος δημοψηφίσματα, ούτε να ζητήσει περαιτέρω μεταφορές αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτείται ομοφωνία και εθνική επικύρωση από όλα τα κοινοβούλια. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν και όπως είπαμε το Εργατικό Κόμμα, ήμασταν ομόφωνοι σε αυτό, εμείς θα είμαστε υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει ο Κάμερον, κάποια μέτρα που θα πάρει μπορεί να μας αρέσουν, εμείς όμως θα στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη για το μέλλον της χώρας. Δεν ήμουν μέλος της οποία αλλά από ό,τι καταλάβα μπορώ να λάβω το λόγο και να μιλήσω. Ειδικά σχετικά με την επιστολή Κάμερον προς τον πρόεδρο του, πρόεδρε, του Συμβουλίου. Θα συνεχίσω στην Ιταλική. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν πολλά αντιφατικά στοιχεία, αν όχι επικίνδυνα, σε με την επιστολή από ε, συνταγματική σκοπιά. Κάποια δεν με εκπλήσουν, μόνο ότι σύμφωνα με τον Ρίτσαρ Κόρμπετ δεν αφορούν opt-out τυπικά αλλά ουσιαστικά πρόκειται για opt-out είναι επικίνδυνο ειδικά το ζήτημα της υποβάθμισης της Ένωσης στο σύνολό της με τις επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα. Κατά να και η, θέση του Μπλεβ ε, διάρκεια της ε, συνθήκης της Λισαβόνας να μην, να μην υλοποιήσουμε μια Ευρώπη διαφορετική αλλά να ε, πειράσουμε την ισχύουσα τονίζοντας τα αρνητικά στοιχεία που η κοινότητα διαθέτει ε, ε, ε, από την σύστασή της. Η Ένωση δεν θα αποτελεί τίποτα παραπάνω από μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών και θα στοχεύει στην ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα που αναφέρεται στο επιστολή. Λοιπόν, όχι η πολιτική Ευρώπη, η οποία αναφέρεται η Mercedes, αλλά ενώπιον ε, μια Ευρώπη η οποία διανύει μια, ε, μια κρίση οικονομική εδώ και χρόνια τώρα, ε, θα περάσω τώρα σε κάποια στοιχεία τα οποία θεωρώ ιδιαίτερα αμφισβητήσιμα. Πρώτα απ' όλα η βούληση να τεθεί η λέξη τέλος με τρόπο νομικά δεσμευτικό στην, ε, ως αφορά την Αγγλία για να δεσμευτεί για μια Ευρώπη όλο και πιο στενά συνδεδεμένη. Σε αυτή τη βούληση συνοδεύονται άλλες δύο επιθυμίες. Η μέγιστη μείωση της κοινή νομοθεσίας που θεωρείται ήδη υπερβολική ε, στα δύο σημεία το Λονδίνο γνωρίζει ότι μπορεί να βασίζεται σε παρόμοιες απόψεις ε, στην Ένωση, ενώ χάρη η κυβέρνηση των κατοχωρών και πολλών, κρατών, πολλών ανατολικών κρατών. Να υπάρξει ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει στα εθνικά κοινοβούλια να ε, αποκλεί κάποιες προτάσεις μη επιθυμητές. Έτσι τα εθνικά κοινοβούλια θα έχουν το δικαίωμα της Πρόκειται για μια εξουσία και αρμοδιότητα που έχει αποκτά ουσία όταν η δημοκρατία και τα κοινωνικά δικαιώματα σε κάποιες χώρες κινδυνεύουν. Σήμερα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως οι πολίτες έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στα εθνικά τους κοινοβούλιο από ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν συμφωνώ, δεν είναι η άποψή μου, αλλά είναι περίπου αυτό το οποίο λέει τόσο το ευρωβαρόμετρο. Άρα δεν ξέρω πώς εμπιστοσύνη μπορώ να έχω σε αυτό. Πάντως το θέμα αυτό μπορεί να αφαιρέσει εξουσίες από το Ευρωκοινοβούλιο, γι' αυτό είναι σοβαρό. Εξάλλου το άρθρο 1 της συνθήκης κάνει αναφορά στους λαούς και στους πολίτες και όχι στα κράτη. Και όταν λέμε πιο στενή ένωση, εννοούμε περισσότερα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο άρθρο 2, που δεν θα πρέπει να έχουν όρια και περιορισμούς βρισκόμαστε ενώπιον της προσπάθειας ε, ελαχιστοποίησης ε, εγγυών που αναγνωρίζονται από τις συνθήκες ανακτώντας ε, περιθώρια εθνικών ελιγμών. Και δυστυχώς αυτό ισχύει ειδικά σε ό,τι φορά το κεφάλαιο περί μετανάστευσης, κλείσιμο των συνόρων απέναντι στα κράτη εκτός Ένωσης, ενεργοποίηση της ε, ελεύθερης κυκλοφορίας μόνο όταν ε, θα υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική σύγκληση, περιορισμός του δικαιώματος στην ελευθερία διακίνησης εντός του ευρωπαϊκού χώρου. Ιδιαίτερα ανησυχητική φαίνεται και η κριτική των ε, δικαστηρίων. Το νομικό opt-out επικρίνεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε ζητήματα μετανάστευσης για λόγους με κατεπίγουσας ε, κρίσης ε, και πριν από την επιστολή Τούσκ, ε, το δικαστήριο του Στασβούργου <clears throat> αναφέρει την απειλή της Αγγλίας αυτή για την έξοδο από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αν δεν γίνουν δεκτές, δεκτά τα αιτήματά της. Και επίσης ο διμερής, η διμερής μέθοδος, η διακυβερνητική που ε, κινδυνεύει να καταλήξει η διαπραγμάτευση. Αυτό που θέλουν να αποφύγουν είναι να υπάρξει μια σοβαρή αντιπαράθεση, σοβαρή συζήτηση με το Ευρωκοινοβούλιο. Και για να κλείσω, εάν μια μεταρρύθμιση της συνθήκης θα πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη μου αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο μέσω της τακτικής διαδικασίας αναθεώρησης ούτως ώστε να συμπεριληφθούν το Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τούτου λεχθέντος θα ήταν επικίνδυνο κατά τη γνώμη μου να ζητήσουμε σήμερα αναθεώρηση των συνθηκών ξεκινώντας από την επιστολή κάμερα για τους λόγους που ανέφερε ο Τζολάιναν. Ο καθένας ε, θα προσπαθήσει να πάρει τα περισσότερα δυνατά πλεονεκτήματα και για τον εαυτό του. Πάντως πιστεύω ότι κάποια στιγμή η συνθήκη θα πρέπει να μετατραπεί και να γίνει σύνταγμα, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η κατάσταση κινδυνεύει να επιδεινωθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Thank you. I also would Ευχαριστώ. Και εγώ πολύ σύντομα θα κάνω κάποια σχόλια. Και εγώ ήμουν αν θέλετε, μέλος της αντιπροσωπείας. Θυμάμαι όμως ε, και την τελευταία θητεία είχαμε επισκεφτεί αρκετές φορές το Λονδίνο. Ήδη φαινόταν ότι θα επανέλθει το θέμα προς συζήτηση, όσον αφορά δηλαδή το θέμα του αν θα μείνει ή αν θα εγκαταλείψει η Μεγάλη Βρετανία το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο ευρύτερα. Αν κοιτάξει κανείς την, την επιστολή συγγνώμη, του Κάμερον, διαπιστώνει ότι πρόκειται ουσιαστικά για πολιτικά θέματα που αφορούν την ε, Μεγάλη Βρετανία και τα οποία συνδέονται με την ευρωπαϊκή πολιτική. Εμείς Σαφώς δεν ξέρω γιατί θα πρέπει να μπούμε στην εσωτερική του συζήτηση για τα δικά τους θέματα σε σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτική. Κάποιες χώρες, αν θέλετε όπως το Ηνωμένο Βασίλειο το θέμα αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Σε άλλες όμως χώρες υπάρχει το θέμα, απλώς έχει μικρότερη διάσταση. Το θέμα είναι πώς έχει προχωρήσει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πώς την καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες αν κατανοούν, αν έχουν εμπιστοσύνη στο, στην Ευρώπη, αν βλέπουν προοπτικές και όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πολιτικά δικαιώματα για θέματα κλιματικής αλλαγής κλπ. κλπ από οικονομικά έως κοινωνικά και άλλα θέματα που αφορούν την πολιτική των κρατών μας. Εμείς λοιπόν, σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σαν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των πολιτών, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αποκτήσουμε κοινέ, ε, αν θέλετε, θέσεις ουσιαστικά πρόκειται για ένα εθνικό θέμα. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να δημιουργήσουμε ε, κίνητρα για την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και δεν είναι δυνατόν με μια επιστολή αν θέλετε να μας απασχολήσει με άλλο τρόπο. Εμείς σαν ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα συζητήσαμε και σήμερα το μεσημέρι αυτό το θέμα. Πώς δηλαδή ερμηνεύουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο θα υπάρξει σαφώς ε, ένα κενό. Ολοκληρώνω. Η συζήτηση αυτή, αν συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά εμείς είναι σαν να οπισθοχωρούμε. Θα πρέπει να είμαστε πιο δυναμικοί, πιο επιθετικοί. Και όπως είπε και ο Τζο και η Μπάρμπαρα, πρέπει σαφώς να πούμε ότι ναι, πρέπει να υπάρξει αλλαγή της συνθήκης, πρέπει όμως να προετοιμάσουμε αυτές τις αλλαγές. Όχι με τον τρόπο που το κάνουμε τώρα, να καταλάβουμε τους φόβους των Ευρωπαίων πολιτών και να βρούμε τρόπους να προσαρμόσουμε αυτά που συμβαίνουν με τις επιθυμίες και την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να πάμε. Να είμαστε λοιπόν προετοιμασμένοι γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να έχουμε αρνητικά αποτελέσματα, όχι μόνο μετά το δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και αλλού. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος... Πάνη ε, Przewodnicząca, Szanowni Państwo, e, bardzo krótko chcę... Mm, Σας ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Jeśli Parlament Europejski ma odegrać rolę e, rzeczywiście jak να πω ότι αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πράγματι θέλει να παίξει ένα δραστήριο ρόλο στη διαδικασία αυτή, τότε πρώτον θα πρέπει να απομακρυνθεί από υπερσυγκεντρωτικές και πατερναλιστικές αντιλήψεις και να υπάρξει περισσότερη κατανόηση, περισσότερη ευαισθησία. Αυτά που είπε ο Κόρμπετ με έπεισαν εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να δώσετε μεγαλύτερο βάρος στις προτάσεις των συντηρητικών, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να μας ενθαρρύνετε να εξετάσουμε με σωστό τρόπο τις τέσσερις προτάσεις κάμερων χωρίς προκαταλήψεις. Και αν υπάρχει η δυνατότητα συμβιβαστική στο εσωτερικό της συνθήκης, τότε ίσως ε, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μιας και βλέπω ότι υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα σε ένα τμήμα των προτάσεων κάμερων και στην έκθεση η οποία προετοιμάζεται από την Επιτροπή μας. Αναφέρομαι στην πρόταση Μπρεσομπρόκ. Υπάρχει, πιστεύω, τρόπος να ανταποκριθεί κανείς με σωστό τρόπο στην ιδέα της κόκκινης κάρτας. Ίσως να, επιβληθεί μια μορφή αυτοπεριορισμού της Επιτροπής ή του Συμβουλίου, όπως είπε ο κύριος Μπρόκ. Ίσως να υπάρχουν κάποια ανώτατα όρια. Αλλά αν τυχόν αποφασίσουμε να υπάρξει η κόκκινη κάρτα, αποφασισουμε να υπαρξει κοκκινη καρτα αυτο δεν σημαίνει ότι θα παραλύσουν τα ευρωπαϊκά όργανα. Αντίθετα, η εντολή θα καταστεί ισχυρότερη και θα μπορέσουμε να τομοθετήσουμε ορθότερα. Πιθανότητες υπάρχουν, δυνατότητες υπάρχουν. Να απαντήσουμε θετικά στα αιτήματα Κάμερον. Επανέρχομαι στο θέμα της εντολής και της νομιμοποίησης. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε περισσότερο ανταγωνισμό ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο γύρω από τα θέματα της εντολής τους. Πολλοί από εσά είπατε ότι εμείς είμαστε εκπρόσωποι 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων και το Συμβούλιο αντιπροσωπεύει με διαφορετικό τρόπο ε, και μάλιστα υπάρχουν και διαφορές ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο εκλέγονται οι κυβερνήσεις Ιταλία, Ολλανδία κτλ. Νομίζω ότι τέτοιε συγκρίσει δεν έχουν νόημα. Ας προσπαθήσουμε όλοι από κοινού να συνεργαστούμε και να βρούμε κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις, ενθαρρύνοντας το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει στην Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλους ομιλητές. Να κάνω και εγώ ορισμένα σχόλια συμπληρωματικά αυτών που ακούστηκαν ήδη και για το ταξίδι και για το θέμα γενικότερα. Ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία περίσκεψης για το τι μπορεί να συμβεί στα πλαίσια της πρώτης επιστολής Κάμερον προς Τούσκ και τι γίνεται ακριβώς με τη διάσκεψη των Προέδρων. Κάποιοι από τους συναδέλφους αντικατέστησαν τους ηγέτες των πολιτικών ομάδων στις συζητήσεις που προηγήθηκαν στο Κοινοβούλιο και δεν είναι σαφές αν το Κοινοβούλιο μπορεί να πάρει μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Ίσως είναι διαπραγματεύσεις στις οποίες δεν ανήκουμε και ίσως η τελική πρόταση να διαφοροποιηθεί εφόσον διατηρούνται τα τέσσερα τα τέσσερα καλάθια ή μάλλον τα τέσσερα στοιχεία του καλαθιού. Περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου και μετά το Κοινοβούλιο θα πάρει πλέον το λόγο γύρω από αυτό. Αντίστοιχα όμως θα θελήσουμε να εμπλακούμε ανάλογα με το είδος ε, του, των μέσων που θα επιλεγούν. Πάντως πολιτικά σε μας ανήκει να αποφασίσουμε πόσο θέλουμε να προχωρήσουμε και σαν ε, σε ατομικό επίπεδο και σαν αύκο. Το Σεπτέμβριο μετά την πρώτη ακρόαση αποφασίσαμε να πάμε στο Λονδίνο. Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τρόπους εμπλοκής και συμμετοχής στον καθορισμό των μέσων που θα οδηγήσουν στις τελικές αποφάσεις και να συμμεριστώ μαζί σας το ότι εγώ πήγα με πολύ περισσότερες ελπίδες στο Λονδίνο σε όλα τα επίπεδα και επιστρέφω λιγότερο αισιόδοξη. Αλλά παρόλα αυτά πεπισμένη ότι το πολύ σημαντικό πακέτο του Κάμερον θα ληφθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπόψη έτσι ώστε οι πολίτες να ενδιαφερθούν, να νιώσουν ασφαλείς. Είναι σαφές ε, ότι οι Βρετανοί ε, ασκούν πολύ σκληρή κριτική στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τη μεταναστευτική κρίση. Λοιπόν, αν καταφέρουμε να δείξουμε πριν το δημοψήφισμα ότι έστω και στην, ε, στο μεταναστευτικό τομέα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, τότε νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες για συζήτηση. Πάντως υπάρχει και το θέμα της Βρετανικής ταυτότητας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και το είπε ο Χέλμουτ όπως και άλλοι συνάδελφοι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο και να προσπαθήσουμε να μην καθυστερήσουμε Έχουμε μισό χρόνο περίπου, δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη όπως σας είπα, αλλά ο Δεκέμβριος δεν είναι η στιγμή που θα γίνουν οι βασικές επιλογές αλλά ελπίζω ε, μέχρι το Φεβρουάριο να ε, μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Έχουμε λοιπόν αρκετούς μήνες μπροστά μας για να δούμε τι σαν αύκο μπορούμε να κάνουμε, να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου στο εσωτερικό των πολιτικών ομάδων. Οι πολιτικές ομάδες είναι, ζηλεύουν τον τρόπο με τον οποίο θα παρέμβουμε Έχουμε όμως μπροστά μας κόσμο ζητήσαμε από τον κύριο Φόλ να μας ενημερώνει τακτικά για το πού πηγαίνουν οι διαπραγματεύσεις. Είπε ότι θα έρθει τον Ιανουάριο τώρα, να δούμε αν θα έρθει και να δούμε τι άλλες δυνατότητες. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει άλλο θέμα, κλείνω τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Α, όχι, οι Μεσεντές. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βρεθεί μια λύση, μια καλή λύση και να μείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπενθυμίζοντας βέβαια και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προς στιγμή Υπάρχει μια άλλη διακυβερνητική διαδικασία και δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι εμείς ε, συμμετέχουμε στη διαδικασία αυτή. Δεν μπορεί κανένας να αποφύγει τα ευρωπαϊκά όργανα που συμμετέχουν. Θα συζητήσουμε το θέμα και στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών να συζητήσουμε το ποιες είναι οι καλύτερες διαδικασίες τις οποίες θα ακολουθήσουμε και στις οποίες θα πρέπει να είμαστε σωστά παρόντες και να μπορέσουμε με ισχυρό τρόπο να φανούμε πολιτικά. Η ΑΦΚΟ είναι θεμελιώδης η παρουσία της σε θεσμικό επίπεδο, αλλά και η ΙΝΚΟ παίζει ρόλο και η ΕΚΟΝ παίζει ρόλο Έστειλα μια επιστολή στον Σούλτς εδώ και αρκετό καιρό για το θέμα αυτό, χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις. Θα τελειώσουμε λοιπόν με το θέμα αυτό. Το τελευταίο θέμα για σήμερα, ενημέρωση για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με την διοργανική συμφωνία. Αυτή τη στιγμή ο ε, Φερχόφστατ ε, ολοκληρώσει τις προτάσεις του στο τέλος Δεκεμβρίου, θα έλθει να τα παρουσιάσει και στη Γιούρη. Όταν το συζητήσαμε το θέμα αυτό, υπήρχε ένα non-paper εξ ονόματος της ΑΦΚΟ που χρησιμοποιήθηκε αρκετά από τους διαπραγματευτές. Η πρωτοβουλία μετά πέρασε στη διάσκεψη των Προέδρων. Ο πρόεδρος Σούλτς θέλει να προεδρεύσει, στην αρχή είπε ότι θα προεδρεύσει, μετά ζήτησε από το Φερχόσταφ να το κάνει και έτσι προσκαλούνται και οι πρόεδροι των δύο επιτροπών, της Γιούρη και της ΑΦΚΟ, κάθε φορά στη συνάντηση των επιτροπών, των προέδρων συγγνώμη, των επιτροπών, όταν ενημερώνει ο κύριος Φερχόστατ. Οι διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει σε πολιτικό επίπεδο και εδώ ο κύριος Φερχόστατ διαπραγματεύεται με τον Νίκολα Σμίτα από το Λουξεμβούργο και με τον Φραντ Στίμερμανς. Πολλή δουλειά γίνεται επίσης σε τεχνικό επίπεδο, όπου έχουμε εκπροσώπους από τα διάφορα ε, θεσμικά όργανα που ασχολούνται με τα ε, θεσμικά. Έχουν 10 κεφάλαια μέχρι τώρα γίνει αντικείμενο μελέτης. Είχαμε 5 γύρους διαπραγματεύσεων που έχουν ολοκληρωθεί. Κάθε φορά που ο Φερχόστατα αναφέρεται στα θέματα αυτά, φαίνεται ότι δημιουργείται μια καλή ατμόσφαιρα και υπάρχει αρκετή δεκτικότητα ε, στις προτάσεις του Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτό θα συνεχίσει και στις τελευταίες φάσεις της διαπραγμάτευσης. Τα κεφάλαια 7 και 8, το 1 προς 6 έχουν περίπου κλείσει αν θέλετε πολιτικά. Τώρα μιλάμε για το 7 και 8 αυτή την εβδομάδα θα υπάρξει μια συμπληρωματική ε, συνεδρίαση και η τελευταία το Δεκέμβριο. Ο Φερχώσταρ πιστεύει ότι θα μπορέσει να κλείσει την ε, διαπραγμάτευση ε, το Δεκέμβριο σε πολιτικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να, έχουμε, να είμαστε βέβαιοι 100% για το τι συμβαίνει, αλλά σύμφωνα με τους κανόνες, τους διαδικαστιστούς, όπως ξέρετε η ΑΦΚΟ είναι η επιτροπή που είναι αρμόδια για τις οργανικές σχέσεις. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι επίσης και για την εξέταση της ε, διοργανικής συμφωνίας ε, γύρω από το θέμα αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τελειώσουμε με την προσπάθεια αυτή, τότε η ΑΦΚΟ θα, συνάψει ένα ψήφισμα, θα συντάξει συγγνώμη, ένα ψήφισμα, συστήνοντας ε, τις θέσεις τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσει το Κοινοβούλιο και αν τα πράγματα πάνε καλά όπως ε, ελπίζει και εύχεται ο κύριος Φερχόφστατ, αυτό σημαίνει ότι ίσως στο τέλος Φεβρουαρίου να υπάρξει μία συμφωνία με τα αποτελέσματα, με σαφή αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Και έτσι τον μήνα Μάρτιο να το εξετάσουμε προσεκτικά και να μπορέσουμε να περάσουμε σε ψηφοφορία τον μήνα Απρίλιο πλέον στην ΑΦΚΟ. Και έτσι τον Μάιο θα φτάσουμε στην Ολομέλεια. Αλλά αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο. Μετά από τις παρουσιάσεις τις οποίες έκανε ο Φερχώστατη, ίσως τα πράγματα να υπάρξουν ε, και καθυστερήσεις. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα. Όταν ο Γκί έρθει εδώ, δεν είναι βέβαιο πότε θα έρθει, αλλά λέμε όταν έρθει εδώ, τον Ιανουάριο μάλλον, θα μπορέσει να μας δώσει την ολόκληρη εικόνα για τη συμφωνία και θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά σε μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομέρειας. Αυτά, αν δεν υπάρχουν άλλα θέματα, ε, τερματίζεται η συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και το απόγευμα είναι η τελευταία... η συνεδρίαση πριν τις γιορτές. Χρόνια πολλά.